Καλωσορίζω τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Σίλβα Καλτέρα και του δίνω αμέσω το λόγο. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κύριε Επίτροπε, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση όσον αφορά τη χρήση του προπολογισμού 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα αρχίσω με τα κύρια συμπεράσματά της. Το 2011 οι λογαριασμοί αντικατοπτρίζουν νομίζουμε σωστά την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα και τις δράσεις της όσον αφορά τη ρευστότητα για το έτος αυτό. Τα έσοδα και οι υποχρώσεις πληρωμών δεν ε, είχαν πραγματικά σφάλματα. Όμως οι πληρωμές επηρεάζονται από πραγματικά σφάλματα με ένα εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος 3,9% για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Το εκτιμόμενο ποσό σφάλματος για το 2010 ήταν 3,7% παρόμοιο δηλαδή. Για να το πω απλά, το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε πολλά παραδείγματα όσον αφορά τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πετυχαίνουν τους στόχους ή όπου οι δαπάνες δεν γίνονται με το βέλτιστο τρόπο. Το μήνυμά μας δηλαδή φέτος είναι ίδιο με τα προηγούμενα έτη. Και παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί το ποσοστό εκτιμούμενου σφάλματος όσον αφορά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, παρόλα αυτά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να δαπανώνται πιο αποφασιστικά, πιο στοχευμένα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και προγράμματα. Συνολικά, τα ελεκτικά συστήματα που έχει εξετάσει το ελεκτικό συνέδριο είναι εν μέρη μόνο αποτελεσματικά και δεν καταφέρουν να εντοπίσουν και να αποφύγουν και να διορθώσουν σφάλματα. Οι δύο κύριοι τομείς ομάδων πολιτικών, δηλαδή όπου το ποσοστό σφάλματος είναι πιο υψηλό, είναι η ακροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, η αλληλεία και η υγεία, όπου το ποσοστό σφάλματος εκτιμάται 7,7%. Όπως επίσης και ομάδα πολιτικής, περιφερειακή πολιτική ενέργεια και μεταφορές, όπου εκεί το εκτιμόμενο σφάλμα είναι 6%. Στους τομείς αυτούς, όπως επίσης και σε όλους τους τομείς επιμερισμένης διαχείρισης, οι εθνικές αρχές είναι Εκείνε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Όμω το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε πολλές περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη απέτυχαν. Για παράδειγμα, στι περισσότερε συναλλαγέ, στην περιφερειακή πολιτική όπου το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε σφάλματα, υπήρχε στη διάθεση των κρατών μελών η ενημέρωση προκειμένου να εντοπίσουν και να διορθώσουν τουλάχιστον μερικά από τα σφάλματα πριν ζητήσουν αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν τούτου, το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε και αντίστοιχα προβλήματα σε άλλους τομείς που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης και στην ομάδα πολιτικής έρευνα και εσωτερικές πολιτικές, όπου το ελεκτικό συνέδριο εκτίμησε σφάλμα 3%. Το ελεκτικό συνέδριο σημειώνει στην έκθεση αυτή ότι οι Γενικοί Διευθυντές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αναγνωρίσει υψηλό κίνδυνο σφάλματος στην ακροτική ανάπτυξη, τη συνοχή και την έρευνα. Αύξησαν την εκτίμησή τους για τον κίνδυνο παρατυπιών στις δαπάνες από 400 εκατομμύρια ευρώ το 2010 σε 2 δισεκατομμύρια το 2011. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, Υπάρχουν βελτιώσεις όσον αφορά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης προτού η οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούμε να πούμε ότι είναι όπως πρέπει. Πολλά από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει κατά το παρελθόν παραμένουν, αν και σε μικρότερο βαθμό. Στην πραγματικότητα, η μείωση στην εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στο σύνολό της δείχνει ότι η βελτίωση των κανόνων και του σχεδιασμού της δαπάνες για τα προγράμματα από τη μία περίοδο στην επόμενη όντως έχει κάποιο αποτέλεσμα. Και τώρα με νομοθετικές προτάσεις για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο που συζητάμε έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία για να διορθώσουμε την κατάσταση. Για πολλά χρόνια το λεκτικό συνέδριο κλήθηκε μάλλον ζήτησε πιο απλά προγράμματα, πιο σαφείς στόχους που να μπορούν ποσοτικά να ελεγχθούν πιο εύκολα. Η φετινή μας ετήσια έκθεση επιβεβαιώνει το μήνυμα αυτό. Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν για καλύτερους κανόνες όσον αφορά τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσουν να εφαρμοστούν οι κανόνες αυτοί σωστά. Έτσι ο προπολεό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά και να προσφέρει έτσι περισσότερα στου Ευρωπαίου πολίτε. Συγχρόνω, εξετάζοντα τι νομοθετικέ προτάσει για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να δημιουργήσουν νέα ευρωπαϊκά συστήματα, μηχανισμούς και διακανονισμούς διακυβέρνησης σε άλλους τομείς ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, εποπτεία του δημοσιονομικού συστήματος και το συντονισμό των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών. Η επιτυχία των πρωτοβουλίων αυτών θα εξαρτηθεί και από την ε, δημοκρατική νομιμότητα και εφόσον δηλαδή υπάρχει αυτή η δημοκρατική νομιμότητα. Σύμφωνα με το Λεκτικό Συνέδριο, ο κατάλληλος έλεγχος, η εποπτεία όλων των κονδυλίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως. Πρόεδρε, αξιότιμοι προβουλευτές. Τα υγιή δημοσιονομικά είναι κάτι που ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελεκτικό συνέδριο δεσμεύεται να συνεισφέρει όσο καλύτερα μπορεί στις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πετύχει αυτό το σημαντικό στόχο με τη δουλειά μας και με την ετήσια έκθεσή μας που έχουμε την τιμή σήμερα να σας υποβάλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Σεμέτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε Καλτέρα, κύριε Σιγητά, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου δημοσιεύεται μια περίοδο που οι νομοθετικοί και οι δημοσιονομικές αρχές θα καθορίσουν τους πόρους για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η άντληση μαθημάτων από την προτερη διαδικασία απαλλαγών και οι νέοι μηχανισμοί διαχει... προτάθηκαν νέα μέτρα διαχείριση και ελέγχου για τα μελλοντικά προβλήματα. Ο νέο δημοσιονομικό κανονισμό εισάγει σημαντικέ μεταρρυθμίσει και εστιάζεται στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στην απλούστευση. Οι, Ευρω... οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχουν σαν στόχο την ενίσχυση τη λογοδοσία όλων των οικονομικών φορέων των εμπλεκομένων. Και τέλος, μηχανισμός ελέγχου για το πόσο το κόστος ελέγχεται αποτελεσματικά εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Αυτά τα προγράμματα πιθανότατα θα καλύψουν στα δυναμίες και τα σφάλματα τα οποία παρατηρούνται τώρα. Στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου στην Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού Νωρίτερα, τα μέλη του Κοινοβουλίου διερωτήθηκαν τι θα μπορούσαν να κάνουν για να βελτιώσουν έτσι περαιτέρω την κατάσταση θα ήθελα να τονίσω ότι εσείς αυτό το κοινοβούλιο ήδη ουσιαστικά συμβάλλετε σε αυτό το στόχο. Πρώτα απ' όλα η μείωση του σφάλματος από 7,3% του 2006 στο 3,9% το 2011 μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο ποσοστό από την παρακολούθηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του που εφάρμοσε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποδεικνύει πόσο χρήσιμο είναι και τι προστιθέμενη αξία δίνει ο επικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των, ε, της αρχής απαλλαγής. Δεύτερον, οι ουσιαστικέ βελτιώσεις στον έδημο συνομικό κανονισμό θα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν χωρί την πολύ ισχυρή συνεργασία μεταξύ, στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Τρίτον, θα πρέπει να εγκριθούν από τους νομοθέτες και άλλες προτάσεις και προγράμματα υπό διαχείριση. Το Κοινοβούλιο ως αρχή της απαλλαγής και συνομοθέτηση έχει κρίσιμο ρόλο να διδραματίσει για την πρόθεση της ορθής οικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο που ανέφερα. Το Συμβούλιο μοιράζεται με το Κοινοβούλιο την ευθύνη εφαρμογής νομικού πλαισίου που είναι στέρεο για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο που θα εγγυάται το σεβασμό της ορθής οικονομικής διαχείρισης των ορθών οικονομικών αρχών. Το Συμβούλιο θα εκδώσει και σύσταση προς το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή. Αυτή είναι μοναδική ευκαιρία να δούμε τι μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση των επιδόσεων των προγραμμάτων στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης. Συνεπώς γι' αυτό ζητώ και την παρούσα Προεδρία και τις επόμενες Προεδρίες να οργανώσουν ουσιαστικές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη επ' αυτών των σημαντικών ζητημάτων. Θα ήθελα να περάσω κάποια μηνύματα όσον αφορά την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2011. Καταρχά, πρέπει να πω ότι για πέμπτη συνεχή φορά το ελεκτικό συνέδριο εξέδωσε θετική γνωμοδότηση ανεφορών για του ετήσιου λογαριασμού Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεύτερον, το γενικό επίπεδο σφάλματο για όλε τι πληρωμέ που κατευρύθησαν το 2011 παραμένει σταθερό εν συγκρίση με το 2010, παρόλο που το επίπεδο κινδύνου των συναλλαγών ε, αυξήθηκε το 2011. Τρίτον, ανάληψη υποχρεώσεων και τα έσοδα για όλο τον προπολογισμό δεν έχουν υλικά ασφάλματα, πραγματικά ασφάλματα και το ίδιο και πληρωμέ για εξωτερική ενίσχυση για ε, βοήθεια, ανάπτυξη, διεύρυνση και διοικητικέ δαπάνες. Τέταρτον, μετά την αύξηση των σφαλμάτων, την αύξηση πέθρου, έχει εφαρμοστεί διεξοδικό πρόγραμμα δράση για να εντοπιστούν τα αίτια αυτών των σφαλμάτων με τη βοήθεια των κρατών μελών και να εντοπιστούν οι αδυναμίες ε, κατά τη διάρκεια της ισχύουσης και της μελλοντικής προγραμματικής περίοδου το ποσοστό σφάλματος για εσωτερική πολιτική αυξήθηκε στο 3%. Εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διάφορες περιπτώσεις για να αποφευχθούν βραχυπρόθεσμα παρόμοια προβλήματα. Πλέον μακρυπρόθεσμα, ο ορίζον 2020 απαιτεί περισσότερες απλουστεύσεις και λιγότερα σφάλματα. Τέλος, για την πολιτική συνοχή το ποσοστό του σφάλματος μειώθηκε σημαντικά από 7,7% το 2010 στο 5,1% το 2011. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι ένα σαφέ μήνυμα. Δείχνει ότι περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εστιάσει την εποπτεία της και τη βοήθεια που χορηγεί στους πιο επικίνδυνους τομείς και τέρους και θα εφαρμόσει αυστηρό έλεγχο διαχείριση ε, και διαχείρισης για τα προγράμματα που είναι υπό την επιτήρηση τη. Και τα κάτι μελη όμω θα πρέπει να αυξήσουν τι προσπάθειέ του. Σύμφωνα το λεκτικό συνέδριο, πάνω από 60% των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν για το Περιφερειακό Ταμείο και 76% για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί από τι εθνικέ αρμόδιε αρχέ πριν αποσταλούν οι αξιώσει του προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιθώριο για βελτιώσει είναι σαφέστατο, πράγματι οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα χαλαρώσουν, δεν θα αφιστούν προσπαθειών για να μειώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο σφαλμάτων. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι ενδείκνεται να τεθεί στο σωστό πλαίσιο το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματο, βλέποντας ποιο είναι, ποια είναι η ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πρέπει να τονίσουμε ότι εντοπιστήσεις αδυναμίε από πλευρά ελεκτικού συνεδρίου δεν οδηγούν σε τεράστιε απώλειε ποσών και σε απάτε. Το βλέπουμε αυτό σαφώ, λαμβάνοντα υπόψη την πολιετή διάσταση των διαφόρων προγραμμάτων και τους διαφόρους μηχανισμούς διόρθωσης και πρόληψης των λαθών. Ανέκτησε και διόρθωσε 1,84 δις ευρώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών το 2011. Ακόμα και αν αυτά τα ποσά αφορούν πληρωμές που κατεβλήθησαν σε προηγούμενα έτη, σε οικονομικούς όρους αυτές οι οικονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις είναι το 1,4% των πληρωμών που κατεβλήθησαν το 2011. Αυτό το στοιχείο δεν συμπεριλαμβάνει ακόμα ποσά που ανακτήθησαν ή διορθώθηκαν από τα κράτη-μέλη στον τομέα της συνοχής κατόπιν των δικών τους ελέγχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να συλλέξει πιο αξιόπιστα στοιχεία από τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε του χρόνου να μπορέσει να παρουσιάσει πληρέστερη εικόνα των διορθωτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεω, αλλά και σε εθνικό μετά από παλιές συστάσεις κατά την απαλλαγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε σοβαρές δράσεις για να αποφύγει σφάλματα. Στην συνοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το 2011 να ξεκινήσει 13 διαδικασίες αναστολής και να διακόψει 105 πληρωμές, συνολικό ποσό 2,75 δις ευρώ. Αυτά τα μέσα θα εφαρμόζονται με αυστηρότητα και στο μέλλον. Από το 2014 και πέρα ελπίζουμε ότι θα συμπληρωθούν και από τους μηχανισμούς διορθώσεων που προβλέπονται για όλα τα προγράμματα υπό κοινή διαχείριση. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομίζεται τις ευθύνες της και θα συνεχίσει προσπάθειες για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στο μέλλον προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των φορολογουμένων θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και πρωτοβουλίες για να καλύψει τις αδυναμίες που ενετόπισε το συνέδριο και θα εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με την αρχή απαλλαγή για να πετύχει τις προσδοκόμενες βελτιώσεις. Ο ρόλος των κρατών μελών είναι ουσιαστικός σχετικά με αυτή την προσπάθεια και η δέσμευση που έχουν αναλάβει να υπομισθούν τις ευθύνες και υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης. Όπως προανέφερα, βασίζομαι στην παρούσα και τις επόμενες προεδρίες να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Δίνω το λόγο στους αγορητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων ξεκινώντας με το ΕΛΚ. Το λόγο έχει ο κύριος Πίπερ για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Παρόλες τις προόδους, ε, η ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, βλέπει, ε, αποδεικνύει ότι αυξάνεται το ποσοστό λάθους για το δεύτερο κατά σειράν έτος και υπάρχουν προβλήματα στο Ταμείο Συνοχής και στην ε, χρηματοδότηση της Υπέθρου. Ε, διαπιστώνω ότι ορισμένα από τα λάθη που διαπίστωσε το ελεκτικό συνέδριο έπρεπε να έχουν διαπιστωθεί από τα κράτη-μέλη και το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Και βεβαίως ε, το ελεκτικό συνέδριο συνεχίζει να αρνείται να δημοσιεύσει και να κοινοποιήσει στα κράτη-μέλη τα λάθη αυτά. Θα πρέπει ε, να υπάρχει μία πιο συλλογική διαχείριση των πόρων και η ερεσιμότητα στα διαρθρωτικά ε, ταμεία πρέπει να υπάρξει μόνο όταν ε, εφαρμόζεται η νομοθεσία και μόνο τότε πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό των ε, σφαλμάτων δεν θα έπρεπε να αναφερθούν σε ποια κράτη αναφέρονται ιδίω όταν έχουν υπάρξει αυτές οι αυξήσεις. Χρειάζεται ένα σαφές μήνυμα και τρίτον το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι απλώς ο διαιτητής μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην ε, νομοθέτηση της γεωργικής πολιτικής πολιτικής ε, και της πολιτικής συνοχής στους μεγάλους αυτούς δημοσιονομικούς χώρους είμαστε οι ρυθμιστές αλλά μπορούμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας διότι υπάρχουν σημαντικές δομές και χρειάζεται ένας ανεξάρτητος δημοσιονομικός έλεγχος από τον Κοινοβούλιο και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στη διαδικασία της απαλλαγής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των σοσιαλιστών ο κύριος Γκάιερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Καλντέρα, κύριε Σεμέτα, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο που υπέβαλε την ετήσια έκθεση που είναι σημαντικό εργαλείο για την διαδικασία απαλλαγής του ε, προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή. Βλέπουμε για 18η φορά ότι υπάρχει μόνο περιορισμένη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως υπεσήμενε και ο κύριος Πίπερ ενώ θέλουμε να υπάρχει μία τάση βελτιώσεως των σφαλμάτων πιο σαφής και δεν δεχόμαστε αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχει και ένα βασικό μήνυμα προς το Συμβούλιο που σήμερα πρόκειται ε, να προσέλθει για να συμβιβαστούμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν περίπλοκες ε, διαδικασίες στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του κοινοτικού προϋπολογισμού θέλει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο δαπανεί ε, τους κοινοτικούς ε, πόρους μπορεί να ξεκινήσει αμέσως και θα έπρεπε ε, να μπορέσουν αμέσως να εφαρμοστούν οι διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, οι κάτω χώρες και ούτω καθεξής. Επίσης είπε ο κύριος Πίπερ ότι σε τομείς σαν την πολιτική ερεύνης διπλασιάζεται το ποσοστό λαθών από 1,4% στο 3%. Πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρεθεί κάποιος τρόπος να μειωθούν και πάλι αυτά τα ποσοστά των σφαλμάτων διότι βλέπουμε ότι είχαμε ποσοστό σφαλμάτων 2% και στο χώρο της υπέτρου έχει αυξηθεί στο 2,7% δηλαδή στην ύπεθρο διαπιστώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων. Ε, πρέπει να ε, δούμε πόσο θα μπορέσουν να καταβάλλονται ε, οι πόροι για την γεωργία. Δεν προσπαθούμε να μην πληρώσουμε αλλά θα έπρεπε ο Επίτροπος Τσόλος να απαιτήσει μαζί με τους συνεργάτες τους καλύτερους ελέγχους για να να μπορέσουμε να πατάξουμε ε, ε, την απάτη και επιπλέον το πρόγραμμα δράσεως του 2008 έχει συμβάλει διότι μπόρεσε να ενισχύσει τους ελέγχους και ο Επίτροπος Σόλος θα πρέπει να προτείνει ε, κάποια λύση για να μειωθεί το ποσοστό των σφαλμάτων. Το ίδιο όμως ισχύει και για την περιφερειακή πολιτική ε, κατά τρόπον ώστε η Γενική Διεύθυνση ε, περιφερειακής πολιτικής να μπορέσει να εμπλέξει περισσότερο την ε, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και θα πρέπει να γίνονται μεταφορές ε, πόρων σε άλλα προγράμματα μόνο όταν έχουν καλυφθεί υποχρεώσεις από τα αρχικά ταμεία. Όταν δεν βρίσκονται τα λάθη θα πρέπει τα χρήματα τα οποία εκκρεμούν να επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των φιλελευθέρων ο κύριος Χατζημαρκάκης για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Καλδέρα, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για τη σημαντική εργασία την οποία εκτελεί κάθε χρόνο προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη και είσαστε η αρχή της απαλλαγής του, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είχαμε ε, συζητήσει πέρυσι την εικόνα της ετησίας εκθέσεων και δυστυχώς η εικόνα δεν έχει αλλάξει πολύ από πέρυσι έως φέτος διότι υπάρχουν πέντε δις που δεν έπρεπε ποτέ να έχουν καταβληθεί ένα ποσοστό σφάλματος 3,9% βλέπουμε ότι υπάρχει μία, δια, μία βελτίωση αλλά όχι και τόσο σημαντική. Πρέπει να δούμε πόσο θα μπορέσουν να αιτιολογηθούν αυτά τα σφάλματα στην Ευρώπη. Επίσης οι δυνατότητες τις οποίες χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο ε, ε, για να προβεί στην απαλλαγή επιτέλους χρησιμοποιούνται και έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στην κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης. Βλέπουμε ότι από το 2008 υπάρχει μία βελτίωση και διακόπτεται τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα που δεν λειτουργούν σωστά. Αλλά πέραν από το ευχολόγιο πρέπει κανείς να δράσει και θέλω να περάσω το μήνυμα και στον Επίτροπο Σεμέτα που σας επιτηρεί. Όσον αφορά την ε, απαλλαγή για τον προϋπολογισμό προϋπολογισμό υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι τα ε, χρήματα τα οποία επληρώθησαν και κατεβλήθησαν χωρίς να υπάρχει δικαίωμα θα πρέπει ε, να επιστραφούν και να λειτουργήσει και αυτή η δυνατότητα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ε, βεβαίως και πολύ σωστά το ελεγκτικό συνέδριο θεώρησε ότι η αξιολόγηση δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική και θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερη η διαδικασία αυτή προς όφελος και του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους πρασίνους. Στάις για 1,5 λεπτό. Κύριε Στάις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι σαφές. Για 8η συνεχή φορά μιλάει για θέμα αξιοπιστίας για το περιθώριο σφάλματος, το οποίο αυξάνει ελαφρά στο 3,9%. Στην γεωργία κυρίως, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στην αλία, στην έρευνα, στην υγεία, στην ενέργεια, στις μεταφορές. Ε, δεν είναι και λίγα. Και κάθε φορά λέει ότι είναι θέμα κακής διαχείρισης και είναι θέμα που προκύπτει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Τα έχουμε τα στοιχεία, 60% διαρθρωτικά ταμεία, στο κοινωνικό ταμείο επίσης. Μα τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να μην υπάρχουν τα σφάλματα αυτά. Οπότε ρωτάω το λεκτικό συνέδριο τι πρέπει να γίνει, δεν θα έπρεπε να πει πιο ξεκάθαρα το λεπτικό συνέδριο ποια χώρα φταίει, ποια κάνει καλά τη δουλειά της και ποια δεν την κάνει καλά. Γιατί αυτό θα βοηθούσε πολύ. Γιατί έτσι θα μπορούσαμε να τα βάλουμε και να εποπτεύσουμε ακόμα καλύτερα τις χώρες που δεν τα καταφέρουν καλά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και τέλος, να δώσουμε περισσότερη σημασία στα δικά μας ε, μέσα, στον ε, ΦΠΑ δηλαδή που συλλέγουμε. Πολλά σφάλματα γίνονται εκεί. Ιδιαίτερα σήμερα που είμαστε σε περίοδο κρίση και που πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καταπολεμώντα ε, την απάτη, να δώσουμε μεγάλη σημασία και σε τέτοιου είδου απάτε που γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για το ECR η κυρία Τσεσκόβα για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Εν γέννη, βλέποντας τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου ανησυχώ. Βασικό πρόβλημα είναι το επίπεδο σφαλμάτων όσον αφορά την κατανομή των πόρων τη Ευρωπαϊκή σε επίπεδο κρατών μελών στην κοινή διαχείριση. Δύο τομεί έχουν ανησυχητικό ποσοστό σφάλματο. Θα πρέπει να θετήσουμε ένα καθεστώ τέτοιο που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίζει δυσκολίε που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη και να αντιδρά εγκαίρω. Το 2011 η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε σε πολλού τομεί με παράβαση των κανόνων Υπάρχουν παραδείγματα στην ετήσια έκθεση και τα παραδείγματα ζωγραφίζουν κακή διαχείριση της χρήσης των δημοσίων χρημάτων. Οι αγρότες συλλέγουν περισσότερους πόρους από ότι ε, αντιστοιχούν στην καλλιεργούμενη έκταση, τα μητρώα δεν είναι πάντα ακριβή και ε, και διάφορα χρήματα που δίνονται κοινωνικού σκοπού ε, δεν δίδονται σωστά, δεν δίδονται σωστέ εκτιμήσει. Η κατάρτιση δεν λαμβάνει χώρα όπω θα έπρεπε. Γίνεται υπερεκτίμηση των δαπανών, λείπει τεκμηρίωση, βρίσκουμε πολλά σφάλματα και σε διαγωνισμούς που διεξάγονται σε πολλαπλή συμμόρφωση, η πολλαπλή συμμόρφωση δεν εφαρμόζεται ούτε από δικαιούχους ούτε από τα κράτη-μέλη. Και τίθεται το ερώτημα, μήπως είναι πολύ περίπλοκοι κανόνες, αυτό ισχύει, ή αυτά τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα απροθυμίας εκμάθησης των κανόνων, εφαρμογής των ε, κανόνων ή μήπως λόγω κακών προθέσεων. Σε περιφερειακή πολιτική πάνω από μισές από τις ε, ε, από, τις, ε, από τα προγράμματα εφαρμόστηκαν δεν είχαν σφάλματα. Όμως τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να διαθέσουν τα περισσότερα σφάλματα πριν ζητήσουν αποζημίωση για τις δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ισχύει μόνο για την περιφερειακή πολιτική, αλλά και για άλλες πολιτικές αυτό. Είναι σαφές ότι οι μηχανισμοί ελέγχου σε επίπεδο κρατών μελών αποτυγχάνουν. Πιστεύω ότι οι φορεί των κρατών μελών πρέπει να είναι αποτελεσματικότεροι και να επομιστούν καλύτερα τι ευθύνε του. Αυτό επί μακρόν το συζητούσαμε. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στου περισσότερου τομεί τη ευρωπαϊκή πολιτική ε, είναι μερικώ αποτελεσματικοί, άρα χρειάζονται πιο διαφανεί κανόνε και καλύτερο έλεγχο όλα τα επίπεδα. Πέρα από του επίσημου ελέγχου, πρέπει να γνωρίζουμε πώ μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα τα χρήματα για προγράμματα που έχουν νόημα και πού δίνουμε προστιθέμενη αξία για τον πολίτη, ευρωπαϊκή αξία στα διάφορα έργα. Αυτό πρέπει να ελέγχουμε. Ευχαριστώ ε, για την, ελευθερία, την Ευρώπη της Ελευθερής Δημοκρατίας. Αντρίσεν για μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι 8 ο χρόνος που δεν μπορεί να δοθεί απαλλαγή από το ελεκτικό συνέδριο και 50% των δειγμάτων δείχνουν παρατυπίες. Οι ιδεολογίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνονται. Φταίνε τα κράτη-μέλη. Εκείνα ε, είναι υπεύθυνα για τις παρατυπίες. Όμως οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα χρήματά τους τα πιστεύονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν κάνει τους ελέγχους που πρέπει να κάνει πριν δώσει τα χρήματα στα κράτη-μέλη. Συνέχεια εμείς ε, καταδικάζουμε το γεγονός αυτό. Όπως επίσης το γεγονός ότι δεν πρόκειται πάντα για απάτες. Όταν ε, κάποιος δηλώνει 150 πρόβατα για παράδειγμα και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν έχει κανένα, αυτό είναι απάτη. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τα χρήματα των φορολογούμενων και κατηγορεί τα κράτη-μέλη, γιατί ζητάει περισσότερα χρήματα για να τα δίνει πάντα στις ίδιες και στις άδειες χώρες. Γι' αυτό και θα έπρεπε να έχουμε περικοπές στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτό περιμένουμε. Και δεν βλέπω γιατί καθυστερούμε. Σας ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, Σόντεργαρντ, για 1,5 λεπτό κύριο Σόντεργαρντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και το λεκτικό συνέδριο για την ετήσια αυτή η έκθεση τόσο υψηλής ποιότητας. Δυστυχώς, όπως το ακούσαμε ήδη, για άλλη μια φορά βλέπουμε πως πηγαίνουμε στην ίδια στραβή κατεύθυνση. 2006 με 2009 το ποσοστό σφάλματος στα λογιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε φτάσει 3,7%. Ήταν μια καλή εξέλιξη. Όμως μετά αυξήθηκε το 2010 ήδη και το 2011 3,9. Είναι όμως ενδιαφέρον ε, να δούμε ότι ο αριθμός ασφαλμάτων έχει αυξηθεί πολύ. 33% 2010, 40% 2011. Όταν ε, τα πράγματα πηγαίναν καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε και το θέλει. Εντάξει, όμως είναι προφανές ότι πια γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται κάθε φορά που αυξάνει το ποσοστό σφάλματος. Εδώ και δύο χρόνια είχαμε μία αύξηση δύο χρόνια συνέχεια του ποσοστού σφάλματος. Δεν είναι αποδεκτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ψάχνει έξω από αυτήν από διοπομπαίους τράγους. Γιατί στο κάτω-κάτω η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις δαπάνες που γίνονται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η επόμενη χρονιά θα είναι καθοριστική. Αν για τρίτη χρονιά έχουμε αύξηση του ποσοστού σφάλματος, εμείς οι Ευρωβουλευτές δεν θα μπορούμε πια να να δικαιολογήσουμε αυτή την κατάσταση στους ε, εκλογείς μας. Πρέπει να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε κάθε χρόνο να βρισκόμαστε στο, σταυρό, στο στραβό δρόμο. Σας ευχαριστώ για τους μη γεγραμμένους. Η κυρία Σινκλέρ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Οι εκλογέ μου δεν θα εκπλήσονται που μαθαίνουν ότι τα χρήματα που μαζεύουν τόσο σκληρά και δίνουν σε φόρου ε, τα σκορπούν, τα διασπαθίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια εβδομάδα πολλά κάτι μέλη ε, έχουν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρούν ότι οι υπηρεσίε που παρέχονται αντιστοιχούν τα χρήματα. Λοιπόν, για, βλέπουμε το ελεκτικό συνέδριο ε, δείχνει ότι έκανα πολλά λάθη μια εκλεγμένη εκπρόσωπη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 60% των σπαλμάτων θα μπορούσαν να έχει εντοπιστεί από τα κράτη-μέλη. Όμω είναι πάρα πολλοί κανόνε, είναι πάρα πολλοί περίπλοκε διαδικασίε και αυτό είναι που φταίει. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το διορθώσει αυτό. Δεν κοινοποιούν καν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα άμεσα προβλήματα που διαπιστώνουν. Ένα από τα παραδείγματα των δισεκατομμυρίων που σπαταλώνται ε, στο Λουξεμβούργο είναι τα 700 εκατομμύρια ευρώ για να να εφαρμοστεί κάτω στο δικαίωμα και να μειωθεί διαφθορά στο κοσυφοπέδι. Τα αποτελέσματα είναι φτωχότατα. Και το προσωπικό που είναι εκεί δεν έχει καν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αν πετάει έτσι ε, τα χρήματα του φορολογημένου μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Και τι γίνεται με ευρωπαϊκό κόμματα τι γίνεται με τα δημοσιονομικά, με τη χρηματοδότηση όπως διαφόρων ακραίων δεξιών ε, κομμάτων, όπως κάποι, ε, τι γίνεται με κάποιους ναζί που χρηματοδοτούνται. Ένας συνάδελφός μου μίλησε για εμπιστοσύνη. Ε, ο λαός της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου όλο πιστεύει και λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δημοψήφισμα κατά πόσο θα πρέπει να μείνει ή να βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Ευχαριστώ στους άλλους αγορητές θα δώσω το λόγο, ξεκινώντας από τον Ορτής, τον κύριο Ορτής, για δύο λεπτά. Η κυρία Ορτής δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σταυρακάκης έχει το λόγο. Buenos ε, Καλή σας μέρα, κύριε Πιστεύουμε ότι το ελεγκτικό ε, συνέδριο μετά τα όσα μας παρουσίασε ο Πρόεδρος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα έπρεπε να ξαναδούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ο καθένας ε, στη δουλειά του, βέβαια, η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να βελτιωθούν. Τα κράτη-μέλη έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη βέβαια και πρέπει να κάνουν πολλή δουλειά προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι όσο γίνεται καλύτερα, όπως βέβαια και η συνολική εικόνα που δίνουμε για τις δαπάνες των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρακάκης έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Καλντέιρα για την παρουσίαση τη ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2011. Στο πλαίσιο τη τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η πίεση στα δημόσια οικονομικά σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερη, συνεπώ η αποτελεσματική χρήση του δημόσιου χρήματο είναι πιο σημαντική από ποτέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη έκθεση του Συνεδρίου, το συνδυασμένο ποσοστό σφάλματο για την περιφερειακή πολιτική, τι μεταφορέ, στην ενέργεια, την απασχόληση και τι κοινωνικέ υποθέσει μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2010 από 7,7 σε 5,1%. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανώνται πιο αποτελεσματικά. Αυτό δεν προποθέτει περικοπή στι δαπάνε, αλλά καλύτερο έλεγχο. Οι εθνικέ αρχέ πρέπει να δεσμευτούν για την καλύτερη διαχείριση του κονδυλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο πάνω από 60% των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή τη περιφερειακή πολιτική θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί από τα κράτη μέλη αν είχαν διενεργηθεί κατάλληλοι έλεγχοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούλτερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Συνεδρίου και στον επίτροπο που δεν ήμουν εδώ στην αρχή της συζήτησης, αλλά είχα άλλες ε, ανηλυμένες υποχρώσεις, άλλη συνεδρίαση δυστυχώς. Άκουσα όμως τι είπαν οι συνάδελφοι που είπαν ότι είναι η 8η φορά που έχουμε την ίδια κατάσταση με το ελεκτικό συνέδριο. Πολύ δύσκολα θα καταλάβει βέβαια το κοινό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως ε, για έβδομη φορά θα δώσουμε απαλλαγή στην Επιτροπή. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει ισχυρά επιχειρήματα για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Έχουμε ε, ε, δοκιμάσει διάφορα. Διακοπή πληρωμών, ψηλά πρόστιμα. Παρόλα αυτά δεν τα έχουμε καταφέρει. Αλλά υπάρχει και ένα πράγμα που δεν έχουμε δοκιμάσει, ενώ το ζητάμε ξανά και ξανά, και είναι ότι όταν δίνουμε λεφτά στις χώρες μέλη να φροντίσουμε να τους δώσουμε να αναλάβουν και μεγαλύτερη ευθύνη και οι χώρες που δεν τα καταφέρνουν καλά να είναι υπεύθυνε. Αυτό βέβαια δεν υπάρχει στην ε, ετήσια έκθεση. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως θα γινόταν. Αλλιώς, ίσως χρειάζεται ένας νέος δημοσιονομικός ε, κανονισμός ώστε να τιμωρούνται οι χώρες μέλη. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα και να προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πρόταση ώστε και τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να μπορούν να δώσουν μια ε, θετική δήλωση και τότε θα μπορούν να τιμωρούνται οι χώρες που δεν τα καταφέρνουν καλά και αντίθετα να λέμε μπράβο σε αυτές που τα καταφέρνουν. Σας ευχαριστώ. Βλάζακ για 1,5 λεπτό. Επόμενος αγωρίτης. Κύριος Βλάζακ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Όποιος διαβάσει την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου θα δει ότι κάποιος κάπου κάνει ένα τεράστιο λάθος. Το ποστό σφάλματος είναι υψηλό, πολύ ψηλό δεν υπάρχουν έλεγχοι και τα διάφορα προγράμματα είναι τόσο εσφαλμένα που πολύ συχνά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δίνουν προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Ένας από τους τομείς που αναφέρεται είναι η πολιτική ανάπτυξη πέθρου, όπου μέχρι 50% ε, των προγραμμάτων έχουν σφάλματα. Το πιο συχνό σφάλμα είναι να μην τηρούνται οι κανόνες όσον αφορά τη διοργάνωση διαγωνισμών και η μη επιλεξιμότητα για τις πληρωμές που καταβάλλονται για προγράμματα. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Διότι δεν είναι ότι οι αποδέκτες θέλουν να εξαπατήσουν, είναι μπερδεμένοι, χάνονται στη γραφειοκρατία, χάνονται στο λαβύριθο των δικασιών. Πολύ συχνά έχουν καλή πρόθεση, προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι και μετά μαθαίνουν ότι έκαναν περισσότερα από ό,τι επιτρεπόταν, ότι έκαναν οικονομίες εκεί που δεν έπρεπε ή παραδείγματο χάρη ότι πρέπει να πιστέψουν κάποια χρήματα γιατί κάποια πινακίδα ή κάποια σημαία πρέπει να βάλουν μπροστά δεν είναι, έχει σωστό μέγεθο. Ε, λοιπόν, χρειάζονται αυστηρότερη έλεγχη, μεγαλύτερη ευελιξία και αυστηρότερε κυρώσει. Αυτό λέει το ελεκτικό συνέδριο. Δεν είναι αυτή η καλή λύση. Η μόνη διόρθωση είναι ριζική αναθεώρηση όλων των κανόνων, απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων και περισσότερες συμπράξεις όσον αφορά τα προγράμματα. Από τη στιγμή που θα είναι απλά τα προγράμματα θα μπορούν να υλοποιούνται και θα μπορούμε να τα επεξεργαζόμαστε ή θα ξέρουμε και τι κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άρτογκ για ένα λεπτό. Κύριος Άρτογκ. Ευχαριστώ. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Παίρνουμε, ε, έχει συμβεί να παίρνουν επιδοτήσεις οι χώρες ε, για 150 πρόβατα για παράδειγμα και να αποδεικνύεται μετά ότι δεν έχουν κανένα. Συνεπώ, μπράβο στο ελεγκτικό συνέδριο για αυτά που λέει. Αλλά δυστυχώ πρόκειται για την κορυφή του παγόβονου που για 8η φορά διαπιστώνουμε την ίδια κατάσταση. Ότι φταίνε τα κράτη-μέλη, ότι παίρνουν επιδοτήσει και ότι τελικά δεν ελέγχουμε όπω θα έπρεπε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Naming and shaming λοιπόν. Να λέμε ποιο φταίει με ονόματα. Διότι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλιώς δεν φαίνεται. Έπειτα δεν είμαστε και αποτελεσματικοί τη στιγμή που πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Είναι πράγματα που τα λέμε χρόνια και χρόνια. Επιτέλους πρέπει αυτό να ληφθεί απόψη και από το λεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε ε, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα σήμερα να αποφασίσω να πω τα πράγματα με το όνομά τους εις βάρος του Συμβουλίου που δεν παρίσταται για να μπορέσει να αντιδράσει και επίσης αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κατακρίνει το 96% των σφαλμάτων, το, το μάλλον των στόχων που έχουμε επιτύσσει χωρίς λα, τι έχει γίνει στο θέμα της ανεργίας, ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας μας, ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας εις τον τομέα της απασχόλησης. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα επί των οποίων θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες διότι στην Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να δείξουμε ότι έχουμε ε, ε, επικοδομητική η παρουσία. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει περισσότερο το τι έχουμε κάνει, τι αποτελέσματα έχουμε ε, επιτύχει και τι μπορούμε να παρουσιάσουμε στους ψηφοφόρους και στους πολίτες. Ε, δεν, ε, για πράγματα που δεν γίνονται από τα κράτη, τι γίνεται με την Ευρώπη. Τι γίνεται κύριε Σεμέτα όταν μία στις πέντε πληρωμές είναι εσφαλμένη στη, στα ευρωπαϊκά ταμεία πόσο αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις ε, τις επιπτώσεις της κρίσεως στους εθνικούς προϋπολογισμούς ε, και επίσης ε, πέστε μου πώς μπορείτε στο μέλλον να επηρεάσετε τους κανόνες τι γίνεται με την συμμετοχή εις ταμεία συνοχής των κρατών μελών και τι γίνεται όταν δεν μπορούν στη συνέχεια να ελέγξουν πού καταλήγουν τα χρήματα και κάθε χρόνο βρισκόμαστε στο σημείο όπου λυπούμεθα για τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε να επιδείξουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Βον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν ε, εισηγητής για την έκθεση ΠΙΦ θέλω να χαιρετήσω την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και όπως ελέγχθη το ποσοστό σφάλματος είναι 3,9%. Θα έπρεπε όμως να τονίσουμε και άλλα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη είναι πολύ σημαντικό ότι όπως είπε ε, το ελεκτικό συνέδριο υπάρχει διαφορά μεταξύ του σφάλματος ε, και της απάτης και μόνο 0,2% των πληρωμών ε, υπόκεινται σε απάτες και ε, δεν έχουν αξιολωθεί με τον ίδιο τρόπο οι υπερβολικές πληρωμές ή οι ελλειπείς πληρωμές και υπάρχουν ακόμη και τα λάθη σε έγγραφα που έχουν χαρακτηριστεί ε, σαν λάθη λογιστικά. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει μία βελτιωμένη αξιολόγηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί ε, χρήζει βελτιώσεως και είναι μια βασική λειτουργία την οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Όλοι πρέπει να βελτιωθούμε και το ελεκτικό συνέδριο και το κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη σχετικά με την ε, πολιτική δημοσίων δαπανών με μία αξιολόγηση καλύτερη του κινδύνου, με καλύτερη διαχείριση των πληρωμών. Γενικώ όμως πρέπει να βελτιώσουμε ολόκληρο το σύστημά μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Έρενχάουζερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι γυρίζουμε γύρω-γύρω διότι κάθε χρόνο ακούμε ε, ότι δεν υπάρχει ε, επαρκές ποσοστό αξιοπιστίας και διαπιστώνουμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Μπαρόζο απέτυχε στο στόχο του που είχε θέσει το 2005. Προχωρούμε με πολύ μικρά βήματα και αυτή είναι και η αχίλιος πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η πηγή τόσων τσακωμών τους οποίους διαπιστώνουμε ε, στις Βρυξέλλες σήμερα. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε να υπάρξει μία μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και για τα έσοδα και για τα έξοδα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και για την λήψη ε, των χρημάτων και για την ε, ε, καταβολή και διανομή τους. Πρέπει να υπάρξουν μακροπρόθεσμοι στόχοι, θα πρέπει να υπάρξουν τα σωστά όργανα όπως η δημοσιονομική η φορολόγηση μάλλον των χρηματικών συναλλαγών κατά τρόπον ώστε να μην συζητούμε πλέον για το τι έχει γίνει και να δράσουμε πιο αποτελεσματικά Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είμαστε για άλλη μια φορά μπροστά στο παράδοξο να έχουμε πετύχει τον έλεγχο και να έχουμε προχωρήσει στο 90% χωρίς σφάλμα, αλλά σε άλλους προπολογισμούς πιο περίπλοκους να μην είναι η ίδια κατάσταση. Έχουμε πετύχει λοιπόν ένα σύστημα ελέγχου για ε, τα πιο περίπλοκα θέματα, χάρη στον ε, διάλογο που έχουμε το Ελεκτικό συνέδριο, το βλέπουμε και με την απαλλαγή, όπως το είπα και συνάδελφοι, για άλλη μια φορά όμως βλέπουμε ότι δεν βγαίνουμε από τον φαύλο κύκλο. Πιστεύω ότι φέτος αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο στα σφάλματα των χωρών μελών για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μα το ξέρουμε ότι πράγματα που βγήκαν από την ΚΑΠ και πήγανε στην ανάπτυξη της υπαίθρου έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έπειτα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Όταν δεν εφαρμόζεται σοβαρός έλεγχος και δεν έχουμε τις απαιτήσει που πρέπει να έχουμε, τότε τα κράτη-μέλη ε, έχουν τα αποτελέσματα που βλέπουμε, αλλιώς δεν θα τα είχαν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε καλύτερο έλεγχο των κρατών μελών. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να ελέγξουμε και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους για να δούμε τι κάνουμε. Θα βλέπαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Όσον αφορά τώρα τα σφάλματα της Επιτροπής, αναφερθήκατε σε αυτό κύριε Σεμέτε, το θέμα της έρευνας μας απασχολεί πολύ γιατί αποτελεί έναν από τους πυλώνες για να βγούμε από την κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα το λύσουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Ντόιτ. Θα του δώσω το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Καλντέρα και τους συναδέλφους του του Ελεγκτικού Συνέδριου για αυτή την ετήσια έκθεσή τους είναι μια αφετηρία πολύ σημαντική για τη διαδικασία της απαλλαγής ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες. Αυτό θα να πω καταρχάς. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι ίσως θυμίζει το περίφημο παράδειγμα αν το ποτήρι είναι μεσογεμάτο μισοάδιο. Ένα πράγμα που ενημερωθεί με δύο τρόπους. Εγώ ανήκω σε αυτούς που θα έλεγαν ότι το ποτήρι είναι μισοάδιο όταν μιλάμε για τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι το δεύτερο έτος κατά το οποίο βλέπουμε αύξηση προβλήματα και συνεπώς όσον αφορά την, την αύξηση των σφαλμάτων, του ποσοστού σφαλμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά τα πράγματα σε εκλογή. Για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο αυξάνονται τα σφάλματα. Κρίμα που δεν είναι εδώ το Συμβούλιο ε, όταν συζητάμε τόσο σημαντικό θέμα. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό, ε, λείπει. Λείπει η μόνιμη εκπροσώπησή του και οι εκπρόσωποι της ε, Προεδρίας. Ακούσαμε να αναφέρω ότι 62% των σφαλμάτων θα μπορούσαν να αποφευθεί. Θα μπορούσαν να το είχαν πετύχει σε επίπεδο 100 μελών. Θα έπρεπε να είναι εδώ να το ακούει το Συμβούλιο. Όμως συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι όσο αφορά τη χρήση των ε, ταμείων συνοχής, τάσεις, ε, βλέπουμε τάσεις βελτίωσης. υπήρχε μια μείωση του επίπεδου σφαλμάτων όσον αφορά τη χρήση των πόρων. Και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Τώρα όμως θα ήταν σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι χρειάζεται λιλεγγύη και συνοχή. Καλύτερη χρήση των πόρων ε, συνοχής ε, χρειάζεται. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι είναι στην αίθουσα ο κύριος Γκόλνιτς. Ούτε συνάδελφος Σαρβάμα. Για ένα λεπτό, συνάδελφε Κλέβα, έχετε το λόγο, κυρία Κλέβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι το 60% των σφαλμάτων στην εκτέλεση της περιφερειακής πολιτικής θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό που δεν έγινε. Πρέπει να δοθεί στο μέλλον μεγαλύτερη προσοχή στην προετοιμασία των προγραμμάτων, κάτι που θα δημιουργούσε πραγματικά προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη. Συμφωνώ με εκείνου που είπαν σήμερα ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη εξίσου. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι οι πολιτικέ συνοχή που είναι από τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη και νέες επενδύσεις. Αυτή η πολιτική συνοχής να, έχει, να είναι ισχυρή για την επόμενη επταετία και να υποστηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμεθα επί περικοπών, αλλά επί καλύτερων ελέγχων και καλύτερη διαχείριση από πλευράς των ευρωπαϊκών κρατών μελών των πόρων αυτών. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε ότι έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα απευθύνομαι στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον ευχαριστώ όπως και όλα τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η κυρία Καλιουλάκη είναι μαζί σας, βλέπω. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για το έργο σας και για τη σημασία που δίνετε στους ευρωβουλευτές. Είναι αλήθεια ότι μας προσέχετε πολύ και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο σε μετά, ο οποίος συνεχίζει το ξέρω το έργο του προκατόχου του προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των λογαριασμών μας. Ο συνάδελφο Μπόγκοσλαβ Σόνικ δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ. Έχει άλλε ανελημμένε κοινοβουλευτικέ υποχρεώσει. Ε, λυπάμαι κι εγώ που δεν είναι εδώ το Συμβούλιο επίση, που είναι η Δημοσιονομική Αρχή. Η έκθεση αυτή βέβαια έρχεται πολύ αργά, Πρόεδρε. Ξέρω ότι δεν φταίτε εσεί. Εγώ έχω υποβάλει τροπολογίε στο δημοσιονομικό κανονισμό για να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πριν την 31η Μαρτίου κάθε έτου να υποβάλει του λογαριασμού και την έκθεσή, της να, την έκθεσή του να την έχει νωρίτερα έτοιμη το ελεκτικό συνέδριο για να μπορούμε εμεί πριν το Δεκέμβριο να ψηφίζουμε. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε Νοέμβριο και να μιλάμε ακόμα για ε, τα λογιστικά του 2011 το ελπίζω να τροποποιηθεί πράγματι το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως το ζητάω. Τώρα έχω και κάποιες παρατηρήσεις. Το άρθρο 323 της Συνθήκης λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φροντίζει ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αναρωτιέμαι, το ελεγκτικό συνέδριο δεν θα μπορούσε εδώ να χτυπάει το καβανάκι κινδύνου κάθε φορά που δεν λειτουργεί καλά το οικονομικό σύστημα. Όταν μα λείπουν 9 δισεκατομμύρια και δεν μπορούμε να πληρώνουμε του λογαριασμού μα ε, δεν θα έπρεπε το ελεγκτικό συνέδριο να μα βοηθάει για να ελέγχουμε του λογαριασμού μα περισσότερο. Έπειτα, για την επιμερισμένη διαχείριση. Εντάξει, το θέμα της ανεξαρτησίας των ελεκτικών οργάνων αλλά νομίζω ότι επιμερισμένη διαχείριση που έχει δείξει ότι είναι χρήσιμη να επανεξεταστεί για να δούμε μήπως τελικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε την δικιά μας δημοσιονομική λειτουργία και να καταργήσουμε την επιμερισμένη διαχείριση που κοστίζει ακριβά και που δεν είναι και αρκετά αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Ιβάνοβα. Είχε τρόπο δύο λεπτά κύριε Ιβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε Καλτέρα, Επίτροπε Σεμέτα, κύριε τα αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου και εγώ, όπω και άλλοι συνάδελφοι, καλωσορίσω την ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού που αφορά το έτο 2011. Θα ήθελα συντομία να σχολιάσω κάποιε στοιχείε που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε. Καταρχά, η κοινή διαχείριση. Η έκθεση δηλώνει το ψήφελο ποσοστό ε, προσφαμάτων στην ανάπτυξη υπαίθρου και περιφερειακή πολιτική που είναι στην κοινή διαχείριση. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μηχανισμών, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί θα πρέπει να απομισθούν τι ευθύνε του συμπεριλαμβανομένοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παραπάνω ακόμα και τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, η άμεση διαχείριση 20% των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεων που δεπανώνται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δήλωσε το Ελεκτικό Συνέδριο ότι για έρευνα και εσωτερικέ πολιτικέ αυξήθηκε το ποσοστό σφάλματο από 1,4% 3% το 2011. Όπω και οι συναδελφοί μου και εγώ θα ήμουν περίεργη. Θα ήθελα να μάθω του λόγου για αυτή την αύξηση και ποια μέτρα εξετάζονται για τη διόρθωση καταστάσεω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, η σχέση μεταξύ αποτελεσμάτων και εισρωών. Καταναλωσορίζω το κεφάλαιο 10 τη εκθέσεω που είναι νέο και δείχνει τα αποτελέσματα του προβλησμού τη Ευρωπαϊκή Ενώση και πιστεύω ότι είναι ένα βήμα προ τη κατεύθυνση ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να μετακυθεί από τη συμμόρφωση προ την επίδοση όσον αφορά τα μοντέλα. Ένα μοντέλο που κοιτάει ποια είναι τα επιτευθέντα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε σαφεί δείκτε, βάσει και στόχου, ούτω ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα επιτέγματα αυτών των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το ελεκτικό συνέδριο στην έκθεσή του δηλώνει σαφώ ότι υπάρχει πεδίο για βελτίωση η Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικότατη πρόκληση να κάνει περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Συνεπώ, όλοι μαζί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, όλοι μαζί θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να δαπανούμε το κάθε ευρώ αποτελεσματικότερα, αποδοτικότερα και να πετυχαίνουμε τα μέγιστα αποτελέσματα αυτή τη εποχή λιτότητα. Διότι αυτό περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτε από εμά. Και τέλο, παρακαλώ, επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, εφόσον είναι η τελευταία μου ομιλία στην ε, Ολομέλεια, να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως συναδέλφους στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και τη γραμματεία μας για την έξοχη συνεργασία μας κατά τη διάρκεια των ετών αυτών. Είμαι ευγνώμων για αυτά τα χρόνια που ήταν γεμάτα από ζωηρές δυναμικές συζητήσεις, έμαθα πολλά από αυτές και ελπίζω ότι συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και μπορείτε να βασίσετε σε μένα ότι ο διάλογος με αυτό το Κοινοβούλιο θα είναι βασική προτεραιότητα στο μελλοντικό μου έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ συνάδελφε Ιβανόβα, καλή τύχη. Και τώρα δίνω το λόγο σε αυτό που ζήτησε για τη διαδικασία προσέγγισης προσοχή του Προέδρου, κάτι και ξεκινάμε από τη συνάδελφο, του συνάδελφο Γκαλπέλτ. Τι συνάδελφο. Ευχαριστώ. Μπορούμε να πούμε συνολικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει καλύτερα τα χρήματα από ό,τι στα προηγούμενα έτη και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίζουν από κοινού κάθε χρόνο για τον ετήσιο προϋπολογισμό αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την καλή χρήση των πόρων και εδώ η κατάσταση χρήζει ακόμη βελτιώσεως. Είμαστε μεν σε καλή κατεύθυνση σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση, αλλά πρέπει να βελτιωθεί ακόμη το ποσοστό λάθους όσον αφορά τον τομέα της συνοχής, της γεωργίας και άλλων τομέων όπου διαπιστώνουμε ακόμη παράνομες πληρωμές και ε, σφάλματα. Βεβαίως ε, ε, είναι θέμα της ευθύνης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών αλλά υπάρχει και ένα συστημικό πρόβλημα δηλαδή δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία σε πολλούς τομείς. Συμφωνώ με τον Επίτροπο. Χρειάζεται κάποια απλοποίηση και εάν ο προϋπολογισμός ε, συρρυκνώνεται πρέπει να τον χρησιμοποιούμε καλύτερα και να ελέγχουμε καλύτερα τη χρήση του. Ευχαριστώ.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 Θα ήθελα να ξέρω τι δικαιολογίες ε, προσφέρουν τα κράτη-μέλη για τους ε, λανθασμένους αυτούς λογαριασμούς. Επίσης ε, θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Αν δείτε την ιστοσελίδα του υπευθύνου λέγεται ότι οι λογαριασμοί δεν έχουν ε, ελεγχθεί και ότι έχει ε, πολλές αποδείξεις, ε, αποδείξεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί και ότι τις δίνει στη γυναίκα του να τα κοιτάξει. Μπορείτε να μου πείτε αν κανένα κράτος μέλος έχει ποτέ πει ναι μεν έχασα τις αποδείξεις μου αλλά δεν χάλασε και ο κόσμος. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Σεμέτα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καλέρα, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Η συζήτηση δείχνει ξεκάθαρα ότι η επιμερισμένη διαχείριση αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τη φετινή διαδικασία απαλλαγή. Όμω υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κονδύλια, με την διαχείρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει όλες τις αιτίε και θα φροντίσει να εφαρμόσει τις συστάσεις σας. Το έργο εξάλλου έχει ήδη αρχίσει. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στην έκθεση ετήσιας δραστηριότητας του Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία αντιστοιχεί πλήρως με την αξιολόγηση του, Ευρω... του Ελεκτικού Συνεδρίου. Βάσει αυτής της έκθεσης ε, και οι γενικοί διευθυντές της ε, Άγκρη, της έρευνας και άλλοι γενικοί διευθυντές πρέπει να ετοιμάσουν συγκεκριμένα προγράμματα δράσης για να βελτιώσουν την κατάσταση στους τομείς που είναι δικιά τους ευθύνη. Οι συνάδελφοί μου, ο Επίτροπος Τσόλος, η Επίτροπος η ο Επίτροπος Χάν κλπ. θα συμμετάσχουν και εκείνοι στην διαδικασία απαλλαγής εξηγώντας τις συγκεκριμένες δράσεις αναλαμβάνουν να προωθήσουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους δικούς τους ε, τομείς. Θέλω επίση να επιστήσω την προσοχή σας και σε μία άλλη πτυχή. Κάποιος μίλησε για περίπλοκους κανόνες. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση περίπλοκοι οι κανόνες και όπως είπα και εισαγωγικά, εμείς θέλουμε στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο ακριβώς να απλοποιήσουμε τους κανόνες. Αυτό όμως που είναι πολύ προβληματικό επίσης είναι ότι οι χώρες μέλη εισάγουν ακόμα πιο περίπλοκους κανόνες. Και ένα μεγάλο ποσοστό σφάλματος οφείλεται ακριβώς στους περίπλοκους κανόνες που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να το εκτάξουμε σοβαρό. Ο για παράδειγμα, αναφέρθηκε στους ίδιους πόρους και για τις, ε, στις απάτες που γίνονται σχετικά με αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει υπόψη της αυτό το πρόβλημα και φροντίζουμε να το λύσουμε. Πιστεύουμε πως τελικά το Συμβούλιο θα εγκρίνει τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει εμείς από αυτού, ώστε να, μειώσει, να μειωθεί πραγματικά το ποσοστό σφάλματος σε σχέση με τον ε, ε, ΦΠΑ και θα φροντίσουμε επίσης και για παρετέρω βελτιώσεις στον τομέα αυτό. Τα μέτρα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί συνολικά η κατάσταση όσον αφορά την συλλογή των ε, ιδιών πόρων. Τώρα υπάρχουν ε, και οι καθαρές βελτιώσεις. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η νομοθεσία που διαθέτουμε σήμερα να συμπεριλαμβάνει και αυτές τις καθαρές διορθώσεις για τη νέα δημοσιονομική περίοδο. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πάμε και έτσι θα υιοθετηθεί ε, σχετική ε, διάταξη για αυτό το θέμα. Τώρα, βασιζόμαστε στην δικιά σας στήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ε, απαλλαγής και σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ελπίζουμε ότι όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, απαλλαγή αυτή θα περάσουν από την προσοχή των κρατών μελών επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δίνω το λόγο στον Πρόεδρο Καλτέρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για τα καλά τους λόγια που τα πήθαν σε μένα και σε αυτούς που εργάζονται στο Συνέδριο. Εστέ βέβαιοι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια που καταβάλλεται, που είναι η βασική μας προτεραιότητα, δηλαδή να έχουμε ορθή οικονομική διαχείριση των δημοσιονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου ζητήθηκε να πω κατά πόσο υπάρχουν ε, όταν λείπουν αποδείξεις αν ο μπορεί να δεχτεί την απάντηση και τι έγινε. Καμιά φορά λείπουν οι αποδείξεις και έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα σαν δείτε στην ε, έκθεσή μας. Λέμε ότι λείπει ε, μία απόδειξη και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Δεν δέχεται να ελεγκτής την απάντηση «Ε, και τι έγινε» πρέπει να παίξετε κι εσείς ένα ρόλο για να αντιμετωπιστούν τα υποβόσκοντα αίτια του προβλήματος. Πολλά αξιότιμα μέρη αναφέθηκαν στην ανάγκη βελτιώσεων. Βελτίωση της κατάστασης. Πρέπει να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν όμως στην αρχή της, της περίοδου προγραμματισμού και πού είμαστε σήμερα. Είδαμε ότι υπήρξε βελτίωση. Τι λέει το ελεκτικό συνέδριο όμως, ότι υπάρχει περιθώριο για αποτελεσματικότερο τρόπο χρήσεως των πόρων, πιο εστιασμένο, πιο στοχευμένο τρόπο χρήσης των πόρων. Οι εθνικές αρχές έχουν θεμελιώδη ρόλο να παίξουν σε αυτό. Διότι είναι η πρώτη γραμμή άμυνας όσον αφορά τους πόρους αυτούς. Αν κανείς δημιουργεί περιπλικότητα διότι απευθύνεται σε εθνικές αρχές για την επιλεξιμότητα ίσως τελικά καταλήξει σε 27 ε, διαφορετικούς κανόνες για επιλεξιμότητα. Και αν ισχύει αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Έχουμε χρυσή ευκαιρία τώρα όσον αφορά τους μελλοντικού κανονισμούς για την επόμενη περίοδο πλαίσιο να αντιμετωπίσουμε τα αίτια των προβλημάτων. Διότι υπάρχουν συστήματα που λειτουργούν για με περίοδο. Δεν περιμένουμε τα ποσοστά σφαλμάτων ή τα πιθανά σφάλματα να πάνε από 0 στο 10 ή από 1 στο 100. Υπάρχουν συστήματα. Αν δεν λυθούν τα αίτια, εξακριβωθούν τα αίτια, δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Η σύστασή μας αξιότιμα μέλη είναι σαφής. Καλούμε. Επί μεγάλο χρονικό διάστημα να υπάρχουν απλοί μηχανισμοί για τη χρήση των πόρων να υπάρχουν σαφείς στόχοι και ελεκτικά συστήματα που είναι αποδοτικά στον αφορά το κόστος. Άλλος στόχος, ποιος θα έπρεπε να είναι, να μπορούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανεχθούμε ή όχι το κίνδυνο σφάλματος σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό είναι καθήκον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το 2004 το Ελεκτικό Συνέδριο κάλεσε αυτά τα θεσμικά όργανα να κάνουν αυτό. Εμείς σαν ελεγκτές έχουμε καθήκον να εξετάσουμε τους τομείς κινδύνων. Και δίνουμε σε αυτό προτεραιότητα. Και κάνουμε σαφείς συστάσεις για βελτιώσεις. Αυτό μας, μας έχει ανατεθεί να κάνουμε και αυτό κάνουμε στο μέτρο του δυνατού. Αλλά και κύριε Φόκαν, τα διοικητικά σφάλματα ίσως προκύπτουν και όταν υπάρχουν, δείχνουν ότι υπάρχουν, υπάρχουν προβλήματα σε ένα σύστημα που τελικά θα δημιουργήσουν προβλήματα υλικά αργότερα στην εφαρμογή προγραμμάτων και θέτουν σε κίνδυνο χρήματα. Πράγματι, κυρία Γκρέσλε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούν για να υπάρχουν εξελίξει. Εκεί που υπάρχει κοινή ευθύνη στη διαχείριση. Και κύριο Ντί, σα διαβεβαιώ ότι σημειώνω δεόντως τις προτάσεις σας για το ρόλο μας ε, να είμαστε ένα είδος συναγερμού να επισημαίνουμε λάθη στο Κοινοβούλιο και θα το εξετάσουμε δεόντως αυτό το αίτημα ε, οι συνάδελφοί μου και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Περατώθηκε η συζήτηση. Στην ημερήσια διάταξη τώρα έχουμε την έκθεση Lifefeed που αφορά την ανάθεση κατεξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων